Mesdames, Messieurs, nous allons commencer nos travaux. Διαπιστώνω ότι όλο και περισσότερο δυσκολευόμαστε να ξεκινήσουμε στην ώρα μα. Κρίμα είναι, εξοδεύουμε τα λεφτά του Κοινοβουλίου. Γιατί πληρώνουμε του διερμηνείς επί 15 λεφτά για να μην κάνουν τίποτα. Λοιπόν, για λόγους ευγένειας, από πλευράς Ευρωβουλευτών, αλλά και για να χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, που θα πρέπει κυρίως να ενδιαφέρει τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, όταν λέμε τρει ώρα, θα πρέπει να ξεκινάμε τρει ώρα. Ως συγητές μας είναι εδώ, οι συντονιστές είναι εδώ, τα πιο σημαντικά μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών είναι εδώ. Σας προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είδατε την ημερησία διάταξή μας. Εάν δεν έχετε παρατήρηση, θεωρούμε ότι η ημερήσια διάταξη υιοθετείται, το σχέδιο δηλαδή της ημερήσιας διάταξης υιοθετείται. Δύο. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχετε τον κατάλογο των γλωσσών που είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχει web streaming και ακούγονται οι εργασίες μας μέσω ίντερνετ. Νομίζω ότι υπάρχει άμεση αναμετάδοση, Πράγματι δεν βλέπω το πράσινο φωτάκι της κάμερας. Έπειτα, για το δημοσιονομικό κανονισμό για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, μετά την ψηφοφορία που έγινε στην ε, μεικτή συνεδρίαση που είχαμε με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, οι δύο συνεισηγητέ μα, η κυρία Κρέσλε από την Επιτροπή Προπολογισμών και ο κύριο Ριβελίνη από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, ξεκίνησαν τι διαπραγματεύσει με τη Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου για να υπάρξει μια συμφωνία ήδη από πρώτη ανάγνωση. Αυτό είχαμε ήδη πει την προηγούμενη εβδομάδα. Οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά ούτω ώστε ε, να βάλουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη του τριμέρου διαλόγου τη 11 η Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, ούτω ώστε, αν όλα πάνε καλά, να υποβάλουμε τον κανονισμό σε πρώτη ανάγνωση, σε μία μοναδική λοιπόν ανάγνωση, στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Επίσης, στο Κομπού News διορθώνουμε το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης το σημείο 6. Είναι ένα σημείο που αφορά το θέμα του ΑΕ για την προσαρμογή των πόρων λόγω του διορθωμένου προϋπολογισμού. Ο Ράιμερ Μπέγκε είναι ο εισηγητής και όχι η Μπάρμπαρα Ματέρα. Η Μπάρμπαρα ανέλαβε κάποια θέματα που τα είχε αρχικά ο Ράιμερ, αλλά όχι όλα. Εν πάση περιπτώσει αυτό σημείο, το σημείο δεν θα το συζητήσουμε σήμερα. Αυτά για το σημείο 2 της ανακοινώσεις. Επίσης, το σημείο 3. Η έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης δεν υπάρχουν πρακτικά δεν υπήρξε συνεδρίαση. Προχωράμε. Σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση αυτή τη εβδομάδα. Σήμερα το απόγευμα θα τελειώσουμε ό,τι είχαμε αφήσει εκρεμές από την, ε, από την ψηφοφορία του προπολογισμού του 2011. Ο εισηγητή μας θα μας παρουσιάσει τις ψηφοφορίες που δεν έχουμε ακόμη διεξάγει και αύριο το πρωί θα σας πρότεινα να αλλάξουμε τα ωράρια που προβλέπονται. Δηλαδή, αύριο το πρωί, στις 8.30 το πρωί, θα γίνει η διάσκεψη των Προέδρων των Πολιτικών Ομάδων του Κοινοβουλίου. Αυτή η διάσκεψη έχει βάλει το θέμα του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ημερήσια διάταξη των εργασιών της. Είναι η τρίτη φορά που διάσκεψη των Προέδρων ασχολούνται με το θέμα αυτό. Και για να συμμετάσχουν στις εργασίες τους έχουν καλέσει την ε, Συντόνια και τη Χέλγκα Τρούπελ, τι δύο εισηγήτρε, καθώς και εμένα, με την ιδιότητα του Προέδρου. Η διάσκεψη των Προέδρων μάθαμε ότι θα ήθελε η ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του 2011 να συνδεθεί πολιτικά με το θέμα του μέλλοντος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών μεσοπρόθεσμα. σε ό,τι αφορά τι δαπάνε που επισύρουν αυτέ οι πολιτικέ, δηλαδή λόγω νέων αρμοδιοτήτων τη συνθήκη τη Λισαβόνας, την επικαιροποίηση των ανωτάτων ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών του πολιτού πλαισίου που ισχύει αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα του mid-term review, τη ενδιάμεση αναθεώρηση που έχουμε θέσει κατ' επανάληψη και ιδίω στην τελευταία έκθεση Μπέγκε που ψηφίσαμε στην τελευταία Ολομέλεια και το θέμα των εσόδων με τη συζήτηση που θα γίνει για τους ιδίους πόρους. Η Επιτροπή Προπολογισμών αυτό το θέμα το έχει συζητήσει επί χρόνια. Επομένως, η διάσκεψη των Προέδρων έχει την πρόθεση να εξετάσει πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επ' ευκαιρία της εξέτασης και της ψηφοφορίας του προπολογισμού του 2011 θα μπορούσε να πείσει το Συμβούλιο και όταν λέω Συμβούλιο είναι το Συμβούλιο Υπουργών, ο συνήθι ομιλητή ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μάλλον, που θα πρέπει να δεχτούν να ξεκινήσει η συζήτηση για το μέλλον των, του προπολογισμού της Ένωσης. Είναι πολιτικό και τεχνικό το πρόβλημα. Αύριο το πρωί λοιπόν, από 8.30 με 10, η διάσκεψη των Προέδρων θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό ακριβώς, με τους συζητητές. Τώρα, θα τους ε, πούμε που έχουν φτάσει οι εργασίες μου και θα των τροπολογιών που προτείναμε στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό 2011, προς το παρόν μόνο για τον προϋπολογισμό του 2011 και θα δούμε ποιε είναι οι θέσει οι προσανατολισμοί και ίσω και οι οδηγίες της διάσκεψης των Προέδρων. Εν συνεχεία, αναβάλουμε, ή αναβάλουμε για τι 9 με 10, αντί για 9, 10 Αντί για 9, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε 10 αύριο τις εργασίες της Επιτροπής μας, έτσι. Χρειαζόμαστε μία ώρα για να ενημερώσουμε και κλεισμένων των θυρών τα μέλη της Επιτροπής, όλα τα μέλη της Επιτροπής, αλλά μόνο τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερωθούν και κλεισμένων των θυρών διότι διεμήθη στην διάσκεψη των Προέδρων. Οι εκπρόσωποι των άλλων θεσμικών οργάνων και όλοι οι θεατές και όλοι οι ενδιαφερόμενοι ναι, ναι. Ε, η διάσκεψη, η συνεδρία θα ξεκινήσει επίσημα στις 11. Με βάση την ε, ημερήσια διάταξη που μόλις τώρα εγκρίναμε. Και θα κάνουμε και τις τελευταίες ψηφοφορίες αν δεν τις τελειώσουμε όλες τις ψηφοφορίες σήμερα. Αυτά λοιπόν για αύριο. Τώρα, για την υπόλοιπη εβδομάδα τι υπάρχει. Υπάρχει μια νέα συνεδρίαση την πέμπτη το απόγευμα, μετά τη μήνυ ολομέλεια, η παραδοσιακή συνεδρίαση της πέμπτης απόγευμα μετά την μήνυ ολομέλεια. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης θα ψηφίσουμε το σχέδιο ψηφίσματος που θα υποβληθεί στην Ολομέλεια και τις τροπολογίες για τον προϋπολογισμό του 2011. Και για τα νέα μέλη θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο στόχος είναι να εξηγήσουμε στα άλλα θεσμικά όργανα και στην κοινή γνώμη την έννοια των τροπολογιών που θα έχουμε ήδη ψηφίσει. Η προθεσμία για τις τροπολογίες στο σχέδιο ψηφίσματος έλυγε σήμερα το μεσημέρι, αλλά φυσικά πάντα υπάρχει η δυνατότητα οι συγητές μας να παρουσιάσουν συμβιβαστικές τροπολογίες. Και ενδεχομένως για να λάβουν υπόψη αυτά που θα ακουστούν αύριο στη διάσκεψη των Προέδρων και εν συνεχεία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Αυτό είναι το πρόγραμμα της εβδομάδας για τις εργασίες μας. Υπάρχουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Όχι. Πάμε στο σημείο 4 της εμερήσιας διάταξης που είναι το τέλος της εξέτασης του σχεδίου προπολογισμού του 2011, οι τελευταίες ψηφοφορίες που χρειαζόμαστε. Ο εισηγητής μας θα μας πει τι μενού μας προτείνει. Συντονία. Dziękuję panie przewodniczący. Zeszłego tygodnia, tak jak pan... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν όντως ορισμένα εκκρεμή ορισμένα υπόλοιπα ή κατάλοιπα που δεν ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά και ορισμένα άλλα προς αποσαφήνιση που δεν τα είχαμε αποφασίσει την περασμένη εβδομάδα. Στο έγγραφο που σας μοιράστηκε υπαριθμών 4 τμήμα 2 εκεί παρουσιάζονται οι θέσεις του προπολογισμού που πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Θα σας πω σύντομα περί τίνος πρόκειται. Στη σελίδα 2 βλέπετε ότι πρόκειται για την κατηγορία 4, τον τίτλο μάλλον 4 όπου υπήρξε πολιτική συμφωνία την οποία πετύχαμε με μεγάλη δυσκολία για τις περικοπές εκεί στο τμήμα 4 Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν τεχνικός να καταρτήσουμε πίνακα. Υπάρχουν πέντε θέσεις παραπάνω που πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Προτείνω λοιπόν όλες μαζί να τις ψηφίσουμε. Δεύτερον θέμα που πρέπει να δούμε σήμερα. Η τροπολογία μου 3.000, υπαριθμούν 3.000 που αφορά το 1α και είναι τροπολογία που προτείνει περικοπή της θέσης για την ίτερ 45 εκατομμύρια αρχικά επειδή όμως στο τέλος άλλαξε η συμφωνία για τα πειραματικά ή πιλωτικά σχέδια και υπήρξαν νέα στοιχεία, χρειαζόμαστε πρόσθετα 2 εκατομμύρια. Και γι' αυτόν τον λόγο προτείνω να μπει το ποσό ως 47 εκατομμύρια. Επόμενη τροπολογία στη σελίδα 4. 4. Την είχαμε συζητήσει την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είμαστε όλοι έτοιμοι να την ψηφίσουμε. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Είναι οι τροπολογίες της ΕΠΕΞ, Πρόσθετη όρη που, που θέτουμε εμείς ως Κοινοβούλιο για την δημιουργία της υπηρεσίας αυτής και αναγκαιότητα πρόσθετων διαβουλεύσεων. Υπάρχει εδώ ένα μεγάλο απόθεμα 18.600.000 αυτό είναι το συνολικό ποσό για την υπηρεσία αυτή και η άλλη τροπολογία, η άλλη αφορά τη μεταφορά προσωπικού από την Γενική Διεύθυνση Ρελέξ στην υπηρεσία αυτή. Σχεσέξ δηλαδή. Άλλες που δεν είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε γιατί χρειάζεται και άλλη συζήτηση με τους συντονιστές τουλάχιστον είναι ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις για τα πειραματικά επιλοτικά σχέδια. Τα, ποσά, τα σχετικά ποσά εγκρίθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αλλά παραμένει το θέμα των σχολείων, γιατί συχνά τα μη εγκριθέντα σχέδια μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες θέσεις, αλλά αυτό απαιτεί πολύ περισσότερη δουλειά και ελπίζω να καταφέρουμε να πετύχουμε σήμερα μια συνένεση ώστε αύριο να είμαστε σε θέση να δεχτούμε με την, σε ψηφοφορία τον συμβιβασμό αυτό. Αυτά είχα να σας πω. Κάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Θα αρχίσουμε λοιπόν τώρα την ψηφοφορία σύντομα. Πρώτη ψηφοφορία όλες μαζί οι θέσεις του τμήματος 4. Υπάρχει πολιτική συμφωνία νομίζω τον Ραν. Να ρωτήσω κάτι, όχι από αυτού. Σε κάτι άλλο, ίσως να μου ξέφυγε κάτι που είπε η Σιδονία. Γιατί μελούσα εδώ με τους βοηθούς μου. Τα δύο αποθεματικά της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης έχουν ξαναμοιραστεί εδώ πέρα με νέα διατύπωση. Θα επανέλθουμε. Ναι, θα επανέλθουμε, λέει ο πρόεδρος, τη στιγμή της ψηφοφορίας είναι οι συμβιβαστικές τροπολογίες που προτείνω και θα μας πει βεβαίως και ο εισηγητής τι άποψη έχει. Για την ώρα, εάν συμφωνείτε όλοι, όσον αφορά τον πίνακα της κατηγορίας 4, είναι ένας πίνακας που διευκρινίζει γραμμή-γραμμή τις λεπτομέρειες πολιτικής συμφωνίας προηγούμενης εβδομάδας για τις οικονομίες που πρέπει να γίνουν μεταξύ της μπανάνας και του ICI από την άλλη για να μείνουμε εντός της ε, οροφής ε, στην κατηγορία 4. Οπότε ζητάω από την Επιτροπή να συμφωνήσει με αυτή την κατανομή, με αυτή την γραμμή και βλέπω πως ο κύριος Πόρτας ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι την εισηγήτρια. λόγω της έκθεσης που συζητάμε είχα την εντύπωση ότι τα συμπεράσματα δεν ήταν τα ίδια με αυτά που προτείνουμε σήμερα που προτείνονται σήμερα έχω λοιπόν ορισμένες αμφιβολίες ως προς το εξής για το Αφγανιστάν τι βλέπετε ως κατανομή. Νόμιζα ότι είχαμε προτείνει και άλλες περικοπές και δεν τις βλέπω εδώ. Ευχαριστούμε. Κάνε ένα άλλο ερώτημα, απορία. Κυρία εισηγήτρια, μπορείτε να απαντήσετε στον κύριο Πόρτα για την μακροπιστωτική βοήθεια. Λοιπόν, κυρία εισηγήτρια. Κοιτάξτε, σας ξαναλέω περί τίνος πρόκειται. Την περασμένη εβδομάδα καταφέραμε την τελευταία στιγμή να πετύχουμε μια πολιτική συνένεση και εγκρίναμε ορισμένες θέσεις στον προϋπολογισμό που ανταποκρίνονταν σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ τους και το Αφγανιστάν. Αντίθετα, οι πέντε επόμενες θέσεις δεν εγκρίθηκαν, δεν ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα γιατί δεν τις ε, έδειχνε ο πίνακας που δεν υπήρχε τότε. Και γι' αυτό σήμερα ψηφίζουμε πέντε πρόσθετες θέσεις. Δεν ξαναψηφίζουμε ό,τι είχαμε εγκρίνει την προηγούμενη φορά. Είναι καινούριε θέσεις. Μάλιστα, τα κατάλαβε και ο κύριος Πόρτας. Λοιπόν, μήπως τότε μπορούμε να ψηφίσουμε τον πίνακα για την κατηγορία 4 στη σελίδα 2. Στη σελίδα 2. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Και εσάς σας ευχαριστώ. αποχέ. Ευχαριστώ και πάλι. Συγχαίρω την εισηγήτρια και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί της. Επρόκειτο για τη δυσκολότερη από όλες τις κατηγορίες για μας και εγκρίθηκε ομόφωνα συγκινητικό. Λοιπόν, με το ίδιο πνεύμα συνένεση συνεχίζουμε για τη θέση που αφορά την ίτερ. Ξαναλέω, επειδή είναι δημόσια η συνεδρίαση και αναμεταδίδεται και στο ίντερνετ παρά το ότι δεν έχει ανάψει το φωτάκι. Μπορεί να υπάρχουν εδώ δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι άλλων οργάνων. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η πολιτική μας θέληση δεν είναι να αμφισβητήσουμε το πρόγραμμα ΙΤΕΡ. Η πολιτική μας θέληση είναι να χρηματοδοτήσουμε καταλήλως τις προτεραιότητές μας. Δεν είμαστε πια στην κατηγορία 4 αλλά στην κατηγορία 1α. Σύμφωνα με την ακριβή στιγμή που θα χρειαστεί να κινητοποιηθούν τα ποσά αυτά. Εξάλλου θα ξαναμιλήσουμε επανειλημμένως για την ΙΤΕΡ και για τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Έχουμε εκεί κάποιο περιθώριο λιγμών. Λοιπόν, η εισηγήτριά μας, σύμφωνα με όσα είχαν αποφασιστεί την περασμένη εβδομάδα, αποσαφήνισε ποια ήταν ακριβώς τα ποσά που χρειαζόμαστε για τη θέση αυτή για να χρηματοδοτήσουμε τις προτεραιότητές μας. Στο έγγραφό σας αναφέρονται 45 εκατομμύρια αλλά μας είπε η συγγήτρια ότι χρειάζονται δύο πρόσθετα εκατομμύρια σύνολο λοιπόν 47 εκατομμύρια 47 στη γλώσσα του Σέξπιρ. Με τα 47 λοιπόν αυτά εκατομμύρια είμαστε κάτω από την οροφή ακόμα. Κρατάμε δηλαδή ένα περιθώριο. Είμαστε ενάρετοι. Και από αυτού λοιπόν τα 47 εκατομμύρια ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Ευχαριστώ. Ποιες; Μία. Δύο. Δύο αποχές. Η θέση αυτή λοιπόν εγκρίνεται. Τώρα η Χέλγα. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Ίσως να καθυστέρησα, ίσως να μην με είδατε, αλλά θέλω να πω μία φράση. Ψήφισα υπέρ της μείωσης αυτής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς ως πράσινοι είμαστε τελείως ικανοποιημένοι από αυτή τη συμφωνία. Δεν καταψηφίζω μεν, αλλά έχω τελείως διαφορετική θέση από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες διότι νομίζω ότι με το ποσό αυτό δεν θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε τις προτεραιότητες μας. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστούμε Χέλγα. Μας το είχατε ξαναπεί βέβαια, αλλά το ξανασημειώνουμε. Για την ομάδα σας λοιπόν τα 47 αυτά εκατομμύρια δεν είναι maximum αλλά minimum. Έτσι ακριβώς. Α, ωραία. Λοιπόν, Λάσλο Σουριάννα. Θέλω να προσθέσω πως δεν νομίζω πως υπάρχει κάποια ομάδα που είναι ικανοποιημένη με αυτά τα οποία κάνουμε, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ε, πρέπει να κάνουμε συμβασμούς και να είμαστε ευέλικτοι. Οπότε και εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος με πολλά πράγματα, αλλά τα υποστηρίζω να κάνω. Ωραία. Όλοι πήραν θέση για το θέμα της ίτερ. Δεν έχετε άλλη επεξηγήσεις, άλλες επεξηγήσεις ψήφου. Ωραία, περνάμε τότε στις δύο τροπολογίες. Κοινή τροπολογία 1 και 2. για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Να σας πω εν παρόδο ότι πρόκειται για δύο τροπολογίες στη διορθωτική επιστολή που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση και τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Είναι οι μοναδικές τροπολογίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υιοθετήσουμε τροπολογίες τέτοιου τύπου και μόνο τότε, εμέσως, σημαίνει ότι ασχοληθήκαμε με την ε, διορθωτική επιστολή και ότι δεν έχουμε να κάνουμε άλλες τροπολογίες στη διορθωτική αυτή επιστολή. Έτσι, φαίνεται αυτονόητο, αλλά το διευκρινίζω. Αν δεν είχαμε υποβάλει τροπολογίες, θα μπορούσαμε να είχαμε αφήσει εκρεμές το θέμα. Ε, λες και θα μπορούσαμε να είχαμε υπονοήσει ότι δεν ασχοληθήκαμε. Αλλά με αυτές τις δύο τροπολογίες δηλώνουμε ότι ασχοληθήκαμε και έχουμε αυτές τις δύο τροπολογίες ακριβώς. Λοιπόν, για αυτό το θέμα συζητήσαμε, θα σας πω τώρα, συζητήσαμε την εβδομάδα για τη δικτύωση, για την Κομισιόν, ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τμήμα 10. Συζητήσαμε στους συντονιστές στην Επιτροπή Προπολογισμού, είχαμε πολλές ε, επαφές έκτοτε και το θέμα αυτό προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα στην Κομισιόν και στην ύπατη εκπρόσωπο της, ε, εξω, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Εγώ ως πρόεδρος τώρα της ε, Επιτροπής Προϋπολογισμών προσπαθώ να διευκολύνω την εξέβρεση μιας λύσης. Δηλαδή, την εξέβρεση μιας διατύπωσης που θα ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουν οι συνάδελφοί μας της ε, Επιτροπή ΑΦΕΤ, τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Μας το είπε και ο πρόεδρο μέσω επιστολής ναι. και τι θεμητέ ανησυχίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΥΠΑ της Ακπροσώπου στα πλαίσια τη άσκηση των αρμοδιοτήτων του όπω προβλέπουν οι συνθήκες. Ναι. Για να τα παντρέψουμε όλα αυτά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και τι δεσμεύσει που λάβαμε στα πλαίσια του τραμερού διαλόγου στη Μαδρίτη τον περασμένο Ιούλιο, τη στιγμή που επιτεύχθη η συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου, Κομισιών, τη ΥΠΑ Εκπροσώπου και του Συμβουλίου για το καθεστώς και τον τρόπο λειτουργίας και τη σχέση με κάθε θεσμικό όργανο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν προτείνω μία μικρή αλλαγή στη διατύπωση των δύο τροπολογιών. Για ποιο λόγο, για τον κάτωθι λόγο. Έτσι όπως είχαν διατυπωθεί στην αρχή, οι τροπολογίες εμέσως υπονοούν ότι το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα ψήφου για κάποιες ε, μεταφορές, ε, μεταθέσεις αν θέλετε προσωπικού ή για κάποιους διορισμούς. Αυτό αμφισβητείται από τα άλλα θεσμικά όργανα όμως. Προτείνω λοιπόν μία διατύπωση πιο ήπια και να μιλάμε στην τροπολογία μόνο για την ανάγκη από πλευρά των άλλων ε, θεσμικών οργάνων, κομισιών και είπα της εκπροσώπου, να ενημερώνουν πριν λάβουν αποφάσεις για μεταθέσεις ή διορισμούς, να ενημερώνουν λοιπόν εκ των προτέρων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μόνο όταν δοθεί αυτή η πληροφορία, αυτή η ενημέρωση, μπορεί να έρθει η επιφύλαξη. Φυσικά το Κοινοβούλιο είναι ελεύθερο να την άρει, να μην την άρει αυτή την επιφύλαξη. Εξαρτάται από την πληροφορία που θα μας δώσουν. Εγώ λοιπόν σας προτείνω μία πιο ήπια διατύπωση. Νομίζω ότι σεβόμαστε και τις συμφωνίες του τραμερούς διαλόγου και τις ευθύνες του κάθε θεσμικού οργάνου. Ο Γκέραν, για αυτό το σημείο. Νομίζω πως όλοι σέβονται τις προσπάθειες της Προεδρίας για να βρεθεί μια λύση γιατί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο το θέμα και το αντιλαμβανόμαστε, αλλά εξακολουθώ εγώ να έχω ένα πρόβλημα με την διατύπωση. Λάβαμε μια επιστολή σήμερα από τα τρία μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών που διαπραγματεύτηκαν τη συμφωνία, οι κύριοι Μπροκ, Φερχόφστατ και Γκουαλτιέρη. Και πρώτα απ' όλα υπάρχει μια επιφύλαξη. Ε, λένε πως για το πρώτο αποθηματικό, για τις προτεραιότητες τελέχωσης. Εσείς το έχετε αλλάξει και λέτε πως θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, που είναι κάτι διαφορετικό βέβαια από το διάλογο. Και διαβάζοντας την επιστολή εδώ πέρα των τριών κυρίων, ε, μιλάνε για διαβούλευση ακόμα. Οπότε μπορούμε να έχουμε λίγο χρόνο να το ελέγξουμε, μπορούμε να το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια mm. της συνεδρίας των συντονιστών και να ψηφίσουμε αύριο. Γιατί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και πρέπει να το δούμε με τους ειδικού μας εμπειρογνώμονες. Θα με ικανοποιήσω πολύ κάτι τέτοιο. Ε, Εάν οι συντονιστές θέλουν περισσότερο χρόνο για προβληματισμό, επειδή εγώ θέλω να βρεθεί αποδεκτή λύση από όλου. και επειδή δεν πιεζόμαστε τρομερά από το χρόνο, εφόσον πιστεύετε ότι κάποιες ώρες διαβούλευσης μπορούν να σας βοηθήσουν και να είναι υποφελείς, γιατί όχι, προκειμένου να επιτύχουμε τον τελικό συμβιβασμό. Συμφωνώ λοιπόν. Nous Ωραία. Αναβάλουμε την ψηφοφορία για αυτές τις δύο τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Ίσως να το ξανασυντήσουμε το θέμα και στη συνεδρίαση των συντονιστών. You ask for the floor. Uh, as it is postponed, I will uh, remark tomorrow. Έχει αναβληθεί, θα επανέλθω αύριο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε τότε πιο γρήγορα. Υπάρχει τώρα η τροπολογία 2062 της Helga Τρούπελ για το Κοινοβούλιο. Έχεις το λόγο, Helga. Ναι, είναι μια τροπολογία που κατέθεσα εκ μέρους του Προεδρείου. Είναι τεχνική προσαρμογή για το προσωπικό της παραγωγής. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Ερωτήσεις. Ερωτήσεις, Helga, για την τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε. Υπέρ της τροπολογίας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Καμία. Υιοθετείτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις. Θα θυμάστε ότι την περασμένη εβδομάδα ψηφίσαμε τα νούμερα, τα ποσά. Τώρα όμως έχουμε και κάποια σχόλια, τα οποία δεν είναι αμεληταία, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις συγχωνεύσαμε πιλωτικά σχέδια. Αυτό όμως τι σημαίνει ότι στα σχόλια θα πρέπει να εντοπίσουμε πολύ καλά ποια, ποιες δράσεις χρηματοδοτούνται από αυτά τα συγχωνευμένα σχέδια. Και σε ορισμένε περιπτώσεις αντικαταστήσαμε τα πιλωτικά σχέδια από σχόλια για τις γραμμές προϋπολογισμού που είχαμε ήδη ψηφίσει. Την ε, τελική γραπτή διατύπωση δεν την έχουμε, στρέφουμε και προς τον εισηγητή να το επιβεβαιώσει καλό θα ήταν να την έχουμε σήμερα το απόγευμα, τόσο ώστε να ψηφίσουμε αύριο. Αν μπορούμε να ψηφίσουμε τις περισσότερες γραμμές on block και χωριστή ψηφοφορία για κάποιες επιμέρους γραμμές στον προπολογισμό. Εντάξει. Είναι πολιτικά ευαίσθητα όλα αυτά τα θέματα και καλό θα ήταν να τα πούμε στους συντονιστάς για να μην δούμε αύριο ψηφοφορίες κατά τμήματα και να μπορούμε όλα να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Α, κάλλιστα. Θα έχουμε λοιπόν αυτόν τον πίνακα καταρτισμένο πριν λήξει η συγκεντρίασή μας. Τον χρειαζόμαστε για να μπορούν όλοι και όλες να δούμε αν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να το πούμε στις συντονιστές μετά. Λοιπόν και στις συντονίστριες. Αύριο η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Νομίζω τα είπαμε τα προκαταρκτικά. Α, όχι. Αύριο επίσης θα ψηφίσουμε την τροπολογία που αφορά τη δημιουργία μιας θέσης για φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που πρότειναν οι σοσιαλιστές. Νομίζω ότι τέτοιες θέσεις μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες, ιδίως για τη συνέχεια, τον επόμενο προϋπολογισμό λοιπόν, και άρα πρέπει να συνσυζητηθούν μαζί με άλλες τροπολογίες και πρωτοβουλίες. στον κέρα. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Δεν νομίζω να υπάρχει καμία δυσκολία να τα ψηφίσουμε αύριο αυτά. Γιατί καλό είναι να έχουμε πρώτα μάθει τι, θέλουν, τι θέλει η διάσκεψη των προέδρων αν, θέλουν, αν έχουν αποφασίσει κάτι για τους ιδίους φόρους ας πούμε. Ο φόρος λοιπόν η φορολόγηση αυτή των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι καλό αφού θα συζητηθεί εκεί να το ξέρουμε και να τα ψηφίσουμε αύριο. Ναι, ναι, πράγματι είναι πιο φρόνιμο έτσι. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντική τροπολογία αλλά διαφορετική πολύ από τις συνήθεις τροπολογίες του προϋπολογισμού. Άρα θα τη δούμε αύριο. Λοιπόν, το 4 νομίζω έχει εξαντληθεί, έχει Όχι, όχι, ο Γκέραντ έχει κι άλλο. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά είχαμε μια αντίρρηση που δεν είχε ψηφιστεί. Είχε ψηφιστεί! Α, εντάξει, τότε Έκανα λάθος. Νόμιζα ότι για την αστυνομική ακαδημία νόμιζα ότι το, δεν το είχαμε ψηφίσει. Η κυρία εισηγήτρια. Δεν ψηφίσαμε αυτές τις παρατηρήσεις. Θα ήθελα να αποφανθεί ο εισηγητής για το θέμα αυτό. Αν ε, μου δίνετε το λόγο, βεβαίω. Πράγματι ψηφίσαμε. Επίσης είπαμε πως θα συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, εξού και αυτή η επιφύλαξη εδώ πέρα στον προπολογισμό του 2011. Όμως, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια τεχνική προσαρμογή για την διατύπωση αυτή για τους όρους άρσης αυτής της επιφύλαξης. Το διάβασα, ήταν ε, σωστό και ήταν καλύτερο νομίζω από την γενική αυτή επιφύλαξη που είχαμε ήταν κάτι πιο ακριβές και το έδωσα στην ε, γραμματεία της ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού η οποία θα την ε, εισαγάγει. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να ψηφίσουμε για αυτήν εδώ πέρα τη διατύπωση. Για μένα, εγώ τουλάχιστον θεωρούσα ότι είχε λήξει η υπόθεση, δεν ξέρω. Ευχαριστώ, Γιούτα. Καλό θα ήταν να υπάρχει το κείμενο, να μοιραστεί και αν υπάρχει πρόβλημα θα το συζητήσουμε σήμερα στους συντονιστές και θα ξανασυζητήσουμε αύριο. Πάντως υπάρχει πολιτική συμφωνία. Υπάρχει μια διατύπωση, έτσι. Ο Γκέραν και οι υπόλοιποι συγητέ ε, θα εξασφαλίσουμε ότι συμφωνούν με αυτή τη διατύπωση, αλλά δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε, καταρχήν τουλάχιστον, επιπλέον ψηφοφορία. Ωραία. Πάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Αν η εισηγήτριά μας είναι εδώ και έτοιμη, προβλέψαμε ανταλλαγή απόψεων για αυτό το σημείο, για το σημείο 5 δηλαδή. Πρόκειται για τα νέα ντοσιέ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής της Παγκοσμιοποίησης. Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ. Θέλω να προτείνω στους συναδέλφους να προτείνω την περίπτωση της Ιρλανδίας αύριο μαζί με την παρουσίαση των άλλων τεσσάρων ετοιμάτων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, έχουμε πέντε υποθέσεις, θα σας παρουσιάσουμε μαζί, γιατί η περίπτωση της Ιρλανδίας θα παρουσιαστεί ούτως ή άλλως, ανάλογα με το τι θέλουν ε, οι συνάδελφοι σήμερα ή αύριο αλλά θα ψηφιστεί στις 26 Οκτωβρίου. Αύριο όμω, ούτω ή άλλω, θα παρουσιάσω άλλε τέσσερι περιπτώσει που θα ψηφιστούν αύριο. Οπότε θα έλεγα να τα αιμοδοποιήσουμε όλα και να τα, να τα συζητήσουμε αύριο. Αν συμφωνείτε βεβαίω. Ναι, ναι. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν. Αλλά μπορείτε να μα πείτε κάποια εισαγωγικά πράγματα σήμερα για να επιταχύνουμε ψηφοφορία αύριο. Αν είσαστε έτοιμοι. Έχουμε λίγο χρόνο για μια ανταλλαγή απόψεων σήμερα, ενώ αύριο θα έχουμε λιγότερο χρόνο και θα έχουμε και πολύ περισσότερε ψηφοφορίε. Επομένω, αν μπορείτε, Μπάρμπαρα, να μα πείτε δύο πράγματα για το σημείο αυτό. Εντάξει, Πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν την παρουσίαση πέντε νέων αιτήσεων για την κινητοποίηση αυτού του ταμείου. Η πρώτη αίτηση θα ψηφιστεί, όπως σας είπα προηγουμένως, στις 26 Οκτωβρίου και αφορά 850 απολύσεις που έγιναν από την κλαδική εταιρεία SR Technics που αφορά τον τομέα των εναέριων ε, μεταφορών. Προβλέπεται ένα ποσό ε, περίπου 7.450.000 ευρώ. Αν λάβουμε υπόψη μας και τις τροπολογίες που έγιναν την περασμένη εβδομάδα, το κείμενο έχει ενσωματώσει και την προφορική τροπολογία που υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Δηλαδή, η δυνατότητα από πλευράς Κομισιόν να εντοπίσει νέα περιθώρια στην γραμμή του προϋπολογισμού, που δεν θα είναι αυτά που προβλέπονται όμως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να βρεθούν νέα δηλαδή θέματα. Αυτή είναι η τροπολογία που έκανα σε σχέση, με βάση την τροπολογία που που ψηφίσαμε και στην, την πρασμένη εβδομάδα. Επίσης, μια νέα αίτηση για 1.429 πωλήσει που έγιναν σε 23 ισπανικές επιχειρήσεις στην Καταλωνία, στον τομέα των αυτοκινήτων. Μιλάμε περίπου για 2.750.000 ευρώ. Τρίτη περίπτωση, 512 πωλήσει που έγιναν στον τομέα των ημιαγωγών στην ε, Ολλανδική εταιρεία NXP ημιαγωγή. 1.800.000 ε, ευρώ. Τέταρτο αίτημα. Από τη Δανία. και αφορά 951 εργαζόμενους που απολύθηκαν από 45 επιχειρήσεις στο Νόντερλαντ, στον τομέα των εξαρτημάτων αυτοκινήτου. Μιλάμε για 7,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Πέμπτη και τελευταία αίτηση της Πορτογαλίας και αφορά 519 απολύσεις στην εταιρεία Κουιμόντα στον ηλεκτρονικό τομέα. Μιλάμε τώρα για 2.400.000 ευρώ περίπου. Φυσικά, οι τροπολογίες που παρουσιάστηκαν για, για αυτές τις αιτήσει είναι οι ίδιες που συζητήσαμε και ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα. Την πρώτη την είχε παρουσιάσει ο Άλβαρο και Άουγλαν, τη δεύτερη οι σοσιαλιστές Νταρντέν, και Γκράιμεντ, αν λέω σωστά το όνομα. Και η τρίτη, Χάουγκλαντ και Αλβάρο. Αυτές τις τροπολογίες όμως τις συζητήσαμε και τις ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως υπάρχει κανένα σχόλιο. Ο κύριος Χάγκλουντ πρώτα και μετά ο κύριος Πόρτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και την εισηγήτρια που μας κάνει τόσο καλές περιγραφές της κατάστασης. Ξέρετε ότι μερικοί από εμάς τους φιλελεύθερους δεν είναι τελείως ικανοποιημένοι. Δεν είναι μυστικό αυτό, αλλά αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο από όλα είναι ότι θέλουμε να υπάρξει κάποια συνένεση και κοινή θέση, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανησυχητική τάση να μην γνωρίζουμε πού πάνε τα χρήματα, όχι όλα τουλάχιστον. Τώρα βλέπουμε να ζητιέται μεταφορά από το ποσό για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και από την πολιτική της ε, καινοτομίας αλλού. Και αυτό μας ανησυχεί γιατί είχαμε πει προηγουμένως ποια είναι η στρατηγική μας και ποιες είναι οι προτεραιότητες μας και τώρα αλλάζουν αυτά. Γιατί φαίνεται ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι δεν είναι σωστή η χρήση που υπήρξε μέχρι τώρα. Υπάρχουν όμως πολύ σημαντικά ποσά που έχουμε εγκρίνει ήδη στις θέσεις του προϋπολογισμού και ξαφνικά προστίθενται και άλλα ποσά. Από πού έρχονται. Κάτι δεν πάει καλά εδώ στους μηχανισμούς μας. Υπάρχουν υπόλοιπα και εξοικονομήσεις. Καλά, μόνο από αυτές τις θέσεις μπορούν να εξοικονομηθούν ποσά. Και αφού υπάρχουν ποσά που δεν έχουν δαπανηθεί, γιατί δεν δαπανήθηκαν. Δεν πρέπει να συνεχίσουν αυτές οι τάσεις. Μπορεί αυτό να μην είναι ακριβώς το θέμα της πρότασης της κυρίας Ματέρα, αλλά πολιτικά συνδέεται. Και για να πάρουμε αποφάσεις για όλες αυτές τις μεταφορές πρέπει να ξέρουμε γιατί ακριβώς και από πού και με ποιο σκοπό μεταφέρονται όλα αυτά τα χρήματα. Αυτό ανησυχεί πολύ τους φιλελευθέρους, σας το επαναλαμβάνω. Γενικά όμως δεχόμαστε τους χειρισμούς της εισηγητρίας. Βέβαια είναι κυρίως ερώτηση που αφορά την Κομισιόν, αλλά θέλαμε και εμείς να το θέσουμε. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Είναι εξαιρετική αυτή η παρατήρηση. Εξαιρετική. Γιατί πράγματι οι θέσεις αυτές έχουν θεωρηθεί ως πρωτεύουσε για μας, προτεραιότητες. Είχαμε πει ότι θα καταθέσουμε τροπολογίες για να αυξηθούν τα ποσά του χρόνου και απ' την άλλη διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως τα ποσά. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν. Κάποτε πρέπει, αν θέλουμε να διατηρηθεί αυτό το ταμείο, να βρούμε και μόνιμο τρόπο χρηματοδότησής του. Το έχουμε ξαναπεί αυτό κατά την συζήτηση της έκθεσης Πόρτας. Μέχρι τώρα χρηματοδοτείται από εξοικονομήσεις που έχουν γίνει λόγω κακής χρήσης άλλων θέσεων. Είχαμε πει από την αρχή ότι η πιο ενδιαφέρουσα θέση ήταν εκείνη που αφορούσε το κοινωνικό ταμείο. Και μα είχε φανεί περίεργο και αντιφατικό. Το είχε πει και η Επιτροπή Απασχόλησης. Τώρα βλέπουμε ότι ζητούν περισσότερα, μεγαλύτερα ποσά και για τα ταμεία καινοτομίας και θέλουμε να μας πει η Κομισιόν αν μπορεί να μας απαντήσει ήδη από τώρα, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως πρέπει να τεθεί το ερώτημα. Ο κύριος Πόρτας μέγαση δήμων των θεμάτων αυτών. Ναι, αυτά τα πράγματα συζητιούνται συχνά. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ιδίω. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τη συζήτηση αυτή την έχουμε ήδη κάνει, αλλά πάντως υπάρχουν δύο απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Πρώτον, υπάρχουν τμήματα του προπολογισμού που όπου η χρηματοδότηση είναι υπερβολική και άλλα όπου δεν αρκεί. Το πραγματικό λοιπόν πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς που μόλις υπόθηκε. Το Ταμείο πρέπει να έχει δική του χρηματοδότηση αν θέλουμε να λειτουργήσει όπως πρέπει. Και εδώ δεν συμφωνώ καθόλου με τον συνάδελφο Άγγλουντ. Δεύτερον, δεν έχω καμία αντίρρηση για τις πέντε πρόσθετες χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται. Βέβαια τα πράγματα τα γνωρίζω καλύτερα για την Πορτογαλία. Αυτή την εβδομάδα συναντήθηκα με εργαζόμενους της επιχείρησης Κιμόντα της Πορτογαλίας που έχει κάποια καθυστέρηση στη χρηματοδότηση. Αυτή οι, 840, 840 εργαζόμενοι είχε προβλεφθεί να τύχουν κάποια μετεκπαίδευση, πράγμα που δεν έγινε. Υπάρχει μια καθυστέρηση λοιπόν, αλλά δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Φταίμε εμείς. Φταίει το σύστημα και η λειτουργία του. Τέλος, την περασμένη εβδομάδα δεν πήρα μέρος μεν στην ε, ψήφιση του προπολογισμού, αλλά ο λόγος ήταν γιατί ήμουν σε άλλη συνεδρίαση με εκπροσώπους των υποψηφίων διαχείρισης αυτών των ταμείων. Η συνάντηση γινόταν στην Πορτογαλία και επειδή ήμουν εισηγητής έπρεπε να είμαι εκεί για να διαπιστώσω πώς η κάθε χώρα προβλέπει το μέλλον του ταμείου αυτού. Η Κομισιόν είχε υποβάλει, είχε κάνει μια έρευνα στις χώρες μέλη, είχε ρωτήσει μάλλον τις χώρες μέλη πώς βλέπουν το μέλλον του ταμείου, ένα ερωτηματολόγιο που είχε αποσταλεί και στους υποψηφίους και όταν εγκριθεί ο προϋπολογισμός καλό θα ήταν να το συζητήσουμε και αυτό. Το πρότεινε ήδη η Κομισιόν δηλαδή να γίνει καταρχάς μια αξιολόγηση των, ε, περιγραφών αυτών για το μέλλον του Ταμείου. Ναι, ευχαριστούμε συνάδελφε. Καλό είναι και αυτό που είπατε. Τώρα, για τις ψηφοφορίες της περασμένη εβδομάδας πράγματι λείπατε, αλλά προσπαθήσαμε να το λάβουμε υπόψη σας τις απόψεις σας όσο γινόταν. Γιατί ο εισηγητής στα, στις προπαρασκευαστικές δράσεις είχε δεχτεί δύο προγράμματα της ΓΚΟΕ, Δύο. Πράγμα το οποίο δημιούργησε και ζήλιες, να το ξέρετε. Πάντως εγκρίθηκαν, εγκρίθηκαν. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή Κομισιόν θέλει ή μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα Χάγκλουντ. Αν θέλει μπορεί να πει και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απάντηση είναι στο κείμενο που μοιράστηκε στην Επιτροπή σας. Μπροστά μου έχω το έγγραφο που αφορά τις πιστώσεις 13 του 2010, υπαριθμών 13 του 2010, για μια μεταφορά πιστώσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην, στην Παγκοσμιοποίηση. Στο έγγραφο αυτό, στη σελίδα 4, αναφέρουμε τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τη δημοσιονομική θέση 05 Είναι μια γραμμή που χρηματοδοτεί διάφορες δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Με την οικονομική κρίση η κινητοποίηση αυτού του ταμείου μειώθηκε. Και επομένως οι πιστώσεις και η χρησιμοποίηση των πιστώσεων μειώθηκαν. Υπάρχει λοιπόν ε, μία δυνατότητα σε πιστώσεις πληρωμών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρίς να φύγουμε καθόλου τις δραστηριότητες που χρηματοδοτεί αυτή η θέση και που όμως υπήρξαν θύμα, όπως σας είπα, της οικονομικής κρίσης και της μείωσης της δραστηριότητας στα venture capitals. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό που αναφέρθηκε, η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Άκουσα τα σχόλια που έγιναν για αυτό το σημείο. Και θα τα λάβω υπόψη μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Γενικό Διευθυντή. Η Μπάρπαρα θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Η συγκήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημειώνω αυτό που ανέφερε ο κύριος Πόρτας, ότι επαναλαμβάνεται η συζήτηση. Αλήθεια είναι βέβαια, αλλά παρόλα αυτά, εγώ ως υπεύθυνη για αυτό το ταμείο και εκπρόσωπος της ομάδας μου του ΕΛΚ, έχουμε κατ' επανάληψη εξηγήσει πώς ψηφίζουμε. Καταλαβαίνουμε ότι θα αναθεωρηθεί το Ταμείο αυτό στα πλαίσια των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών, όταν γίνουν δηλαδή διαπραγματεύσεις για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Τώρα, αυτή τη συζήτηση θέλουμε να τη συνεχίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμό ή να γίνει αλλού. Ε, υπάρχει και η Επιτροπή Σούρε. Συχνά τα μέλη είναι τα ίδια θέλουμε να συζητήσουμε εδώ στον προπολογισμό ή να τη μεταφέρουμε τη συζήτηση στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ. Όλοι γνωρίζουμε ότι το να βρούμε κάποια ποσά, κάποια περιθώρια για, αυτό το, για αυτή τη δημοσιομική θέση είναι δύσκολη. Κοιτάξτε, μου, φέρνε μου φέρνει στο μυαλό την εικόνα της α, ε, κοντής κουβέρτας. Αν την τραβήξω προς το πρόσωπο ε, εκθέτω στο κρύο τα πόδια μου και αντίστροφα. Αν την τραβήξω προς τα πόδια θα εκθέσω το πρόσωπό μου. Το θέμα είναι να συζητηθεί αυτό το θέμα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης σε μια επιτροπή που, θα, είναι αρμόδια για το μέλλον του. Εδώ θα συζητήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό ή στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ. Το, θέμα αυτό, το, το ερώτημα αυτό το θέτω ε, και θέλω να μου το απαντήσουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή Σούρα θα πρέπει να προτείνει την τελική λύση. Προφανώς. Αλλά μπορεί να χρειαστεί και εμείς να προσαρμόσουμε το μηχανισμό εκ των προτέρων. Εξαρτάται από τον αριθμό των φακέλων και από τα χρήματα που υπάρχουν στη διάθεσή μας. Εάν τη στιγμή που βγαίνουμε από την κρίση ο αριθμό των φακέλων μειώνεται, τότε μπορούμε να περιμένουμε τι εργασίε τη Επιτροπή Σούρε και το μελλοντικό πολιετέ πλαίσιο. Αν όμω, δυστυχώ, ο αριθμό των φακέλων αυξηθεί, αυξηθούν οι αιτήσει και οι πηγέ χρηματοδότηση μειωθούν, γιατί θα ψηφίζουμε προπολογισμού όλο και πιο μικρού, σφιχτού, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμόσουμε το μηχανισμό μας, έτσι, τον τρόπο συζητήσεων. Τον κύριο Νταρντέν τον ξέχασα, δεν τον είδα μου είπανε και ο κύριος Άγγλουντ. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έχω την ε, συνήθεια να κοιτάζω την, α, προς τα άκρα αριστερά. Η Γιούτα βέβαια είναι ακόμα πιο αριστερά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι τυχερός άρα που κάθομαι στο κέντρο και συνέχεια μιλάω. Θέλω να σοβαρευτούμε. Ένα σύντομο σχόλιο. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή που μας διαφώτισε λίγο για την γραμμή αυτή του προϋπολογισμού αλλά το θέμα είναι πως αν δούμε τα πράγματα πριν από λίγες εβδομάδες τα χρήματα δεν έφυγαν από αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού τόσο δεν έχω τα χαρτιά μου τώρα μαζί αλλά εάν το δει ο κύριος Γενικαίος Διευθυντής ε, δει όλες αυτές τις γραμμές θα δει πως είναι όλες από τον ίδιο τομέα και ενδιαφέρον είναι γιατί υπάρχει τμήμα ε, αυτού του προπολογισμού που έχει ε, χρήματα τα οποία περισσεύουν και αυτό ίσως ε, θα μπορούσε να μας εξηγήσει τι γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Ενθαρρύνω λοιπόν την Κομισιόν να το δει, ειδικά όταν ξέρουμε πως τα ιδιωτικά αυτά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου πέρσι μειώθηκαν και Βεβαίω, το να έχουμε εμεί αδιάθετα κονδύλια δείχνει πω υπάρχουν προβλήματα ίσω με του δημοσιονομικού κανονισμού που δεν καθιστούν δυνατή τη χρήση αυτών των χρημάτων εκεί όπου χρειάζεται. Αν ακούσετε τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών, είναι σαφέ πω χρειάζονται λεφτά ακριβώ σε αυτού του τομεί. Οπότε κάτι πάει καλά με τι δομέ μα εδώ πέρα. Και αυτό θα έλεγα να κοιτάξει η Κομισιόν. Ειδικά όταν μιλάμε για πολλές γραμμές του υπερπολογισμού με αδιάθετα κονδύλια. Και... Καλό είναι νομίζω να το κοιτάξει αυτό και η Κομισιόν για του χρόνου, γιατί όπως είπε και ο κύριος Λαμασούρ, θέλουμε περισσότερα χρήματα για του χρόνου, αλλά δεν έχει νόημα να βάζουμε εμείς χρήματα και να μένουν αδιάθετα. Ας κόψουμε τις γραμμές αυτές του προπολογισμού. Το Πρόεδρε, δύο προβληματισμούς για τη μεταφορά κονδυλίων. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Πόρτας. Πόρτας. Σημειώνω και καταγράφω την αντίδραση της κυρίας Ματέρα. Όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό, ε, μιλήσαμε για, την, ε, το πρόβλημα αυτό των μεταφορών. Εμείς ως ομάδα ήμασταν κατά των μεταφορών, γι' αυτό όταν ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα ε, υποβάλαμε τροπολογία. Είμαστε κατά της τεχνικής των μεταφορών. Όποιο και αν είναι το ποσό, όποια και είναι η πίστοση που μεταφέρουμε. Θα πρέπει να είναι σταθερό αυτό το ταμείο, θα πρέπει να έχει την δική του θέση προπολογισμού, θα πρέπει να είναι σταθερή αυτή. Ε, να το συζητήσει και η Επιτροπή Σούρε. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να πρικοδοτήσουμε καλύτερα αυτό το ταμείο. Είναι σημαντικό δεδομένου του αριθμού των αιτήσεων και φοβάμαι ότι δεν θα μειωθούν οι αιτήσει προ αυτό το ταμείο. Δυστυχώ. Αλλά δεν θα μειωθούν. Δεύτερο σχόλιο για την απάντηση που μας έδωσε ο Γενικός Διευθυντής της Κομισιόν. Δεν μας ικανοποιεί αυτή η απάντηση. Ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά δεν είναι παράδοξο τη στιγμή της κρίσης να έχουμε υποπορόφηση ε, των κονδυλίων αυτού του ταμείου. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι πολλές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είχαν ανάγκη από αυτές τις ε, πιστώσεις για τα κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου, τα venture capitals. Ελπίζω να έχουμε την δυνατότητα λοιπόν να επανέλθουμε στο θέμα τη ε, χρήση αυτών των πιστώσεων και να μα δώσει περαιτέρω εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρο, η κρίση έχει ίσω αντιφατικέ επιπτώσει. Γιατί από τη μία υπάρχουν πρόσθετες ανάγκες χρηματοδότησης για τις επιχείρησει, από την άλλη όμω, είναι λιγότερα τα προγράμματα αφού υπάρχει κρίση και οι τράπεζες πάβουν να χρηματοδοτούν επενδύσεις. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από την αγορά την ίδια. Εφόσον όμως εδώ δεν χρηματοδοτούν οι τράπεζες υπάρχει λιγότερη καινοτομία. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει τους τελευταίους μήνες. Ίσως να μην κρατήσουν πολύ καιρό όλα αυτά, αλλά τα ερωτήματα αυτά είναι όντως πολύ σοβαρά και θα πρέπει κάποτε να τα απαντήσουμε. Κυρία Χάουκ, και ως αντιπρόεδρος της Κομπούς και ως πρόεδρος της Επιτροπής Σούρε. Γιούτα η Σοφή θα μας μιλήσει. Ναι, και αυτό το οποίο είπε η Μπάρμπαρα είναι σωστό. Είμαστε στο 2010. Η Επιτροπή αυτή οπωσδήποτε θα μας πει τι, τι θέλει για το εάν θέλουμε να συστήσουμε ένα ταμείο ή αν θα είναι κάτι το εικονικό ή αν θα πάει σε διαφορετικά σημεία του προπολογισμού. Αυτό θα το διαπιστώσουμε τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Αλλά εμείς στην Επιτροπή μας θα πρέπει από το ένα έτος ε, του προπολογισμού στο άλλο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την τωρινή ε, κατάσταση την νομική. Και σωστό είναι βέβαιο ε, αυτό το οποίο είπε ο Καλχάγκλουντ και εγώ νομίζω πως, όπως είπε και ο πρόεδρός μας, ο Αλέν πως πολλές επιχειρήσεις δεν θέλουν να επεκταθούν ούτε καν να ξεκινήσουν δραστηριότητα και το ξέρω αυτό γιατί έρχονται και παραπονιούνται σε μένα οι επιχειρηματίες γιατί οι τράπεζες δεν δίνουν τα λεφτά τα οποία, δεν διοχετεύουν τα λεφτά τα οποία τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή γενικά με την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να υπάρξει ακριβώς αυτή, ε, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα που έχουμε για τον κίνδυνο. Γιατί δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα στον τελικό δικαιούχο. Εκεί πέρα πρέπει να δουλέψει η Κομισιόν και να κάνει κάτι. Ναι. Νομίζω λοιπόν πως... Εντάξει, μπορεί να δίνει το Κοινοβούλιο λεφτά, αλλά εάν δεν φτάνουν τελικά εκεί που θέλουμε δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και ξανά τα ίδια θα λέμε κάθε χρόνο. Οπότε πρέπει να το συζητήσουμε αυτό οπωσδήποτε στην Επιτροπή και πρέπει εμείς ως ε, κοινοβούλιο να τοποθετηθούμε κατά πλειοψηφία, αλλά να δούμε και τι θα κάνουμε με το πώς έχουν τώρα τα πράγματα. Να βρούμε μια λύση με την τωρινή την νομοθεσία για τον προπολογισμό του επόμενου έτους. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση. Κατάφεραν δηλαδή τα κράτη-μέλη να υπάρχει τώρα αυτό το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης για να λάβουν περαιτέρω κονδύλια για τις δραστηριότητε τους και τώρα έχουν τις ε, κατευθυντήριες γραμμές, έμαθαν τις κατευθυντήριες γραμμές οπότε τώρα νομίζω θα έχουμε πιο συχνά αιτήματα. Ευχαριστώ κύριο Σκάβελ. Ευχαριστώ. Έχουμε να κάνουμε με πρόβλημα λόγω συστήματος. Αν είχαμε ένα σύστημα προϋπολογισμού, ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, διαφορετικό, θα, θα δουλεύαμε αλλιώ. Χρειαζόμαστε μια κάποια ευελιξία Το θέμα είναι με αυτά τα δεδομένα πώς μπορούμε να βρούμε τη λύση. Με δεδομένα το σύστημά μας, με δεδομένη την ευελιξία που έχουμε κτλ. Τώρα, για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ίσως και αυτό θα πρέπει να έχει ίδια πρικοδότηση. Αυτό που είπαμε ο Γενικός Διευθυντής είναι αληθές. Οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας είναι συμπληρωματικοί. Αντιμετωπίζουμε τώρα την οικονομική κρίση και, και στη χώρα μου βλέπω ότι οι επιχειρήσεις περιορίζουν τη δραστηριότητά τους. Δεν θέλουν να ξανοιχτούν. Θα έχουμε και λιγότερα προγράμματα από τη μία και από την άλλη θα έχουμε τη δυνατότητα πρικοδότησης του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Η εξήγηση που μας δόθηκε είναι σωστή, είναι λογική και χαίρομαι που έχουμε αυτά τα μέσα. Και όπως και η Γιούτα, και εγώ θα ήθελα αυτό το ταμείο να χρησιμοποιηθεί για την καινοτομία, αλλά προς το παρόν δεν είναι δυνατόν. Πρόεδρος, σωστό είναι αυτό, γιατί σε περίοδο κρίσης, αν δεν υπάρχει άμεση προοπτική νέων αγορών, είναι επικίνδυνο για μια επιχείρηση να ξεκινήσει νέες δραστηριότητε. Αν δεν υπάρχουν πελάτες, ας πούμε, τώρα αμέσως, τι γίνεται. Δεν έχει νόημα να ανοιχτεί. Τώρα, για τις ε, δημοσιονομικές ε, γραμμές που υπάρχει λόγω της αρχής της ε, προσθετικότητας, συγχρηματοδότηση. Ο, το, το δημόσιο των κρατών μελών που είναι τέρος, ας πούμε, δεν έχουν πόρους να συγχρηματοδοτήσουν. Τώρα, για να κάνω μια σύγκριση στον τομέα της, με τον τομέα της πολιτικής υγείας. Όταν υπάρχει μια επιδημία γρήπης, αφιερώνουμε πολύ περισσότερα χρήματα ε, στους ε, αρρώστους παρά στην προετοιμασία των πρωταθλητών για τους Ολυμπιακούς. Επομένως, λογικό είναι όταν δεν υπάρχει επιδημία να δίνουμε και λεφτά για να προετοιμάσουμε και τους πρωταθλητές παρά να δίνουμε λεφτά εφόσον δεν υπάρχουν ασθενείς σε υποθετικούς ασθενείς. Ευχαριστώ. Εγώ ικανοποιήθηκα πάρα πολύ με τις ε, παρατηρήσεις ε, του κυρίου Χάγλουντ και συμφωνώ, αλλά νομίζω πως και εμείς θα πρέπει να δούμε το τι γίνεται με το εξή. Μεγάλες επιχειρήσεις ζητάνε κάλυψη από το Ταμείο, αλλά οι μικρές και οι μεσαίες όχι. Οπότε η Κομισιόν θα πρέπει είτε να απλοποιήσει και να επιταχύνει την διαδικασία για να ξέρουν πού βρίσκονται οι επιχειρήσεις, είτε να μοιράσει τα χρήματα αυτά στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν αυτά μετά να τα διαθέσουν σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Μπορεί να κλείσει λοιπόν η ανταλλαγή απόψεων για αυτό το σημείο. Υπενθυμίζουμε ότι για το Ιρλανδικό αίτημα, στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, προβλέπεται ότι η γνωμοδότηση θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης 26 Οκτωβρίου και εμείς θα ψηφίσουμε στην Κομπή την ίδια ημέρα, ούτω ώστε να περάσει στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου το σημείο αυτό, το 5 για την Ιρλανδία. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αιτήματα της Πορτογαλίας, το αίτημα της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Δανίας, σημεία 8, 9, 10 και 11 της Μέσιας Διάταξης, η Επιτροπή Απασχόλησης γνωμοδότησε στις 30 Σεπτεμβρίου για τα τέσσερα αυτά θέματα και εμείς θα ψηφίσουμε αύριο. Εισηγήτρια. Ναι, σωστά τα είπατε. Μόνο μια μικρή διόρθωση η επισήμαση. Να υπενθυμίσω στου συναδέλφου ότι σε ό,τι αφορά το Ιρλανδικό αίτημα υπάρχει δυνατότητα να παρουσιαστούν τροπολογίε μέχρι τι 20 Οκτωβρίου. Έτσι. Μόνο αυτό να το ξέρουν οι συνάδελφοι, μια και υπήρχε ενδιαφέρον ε, για τη συζήτηση. Μπορεί να υπάρξουν λοιπόν και νέε τροπολογίε μετά από αυτό το έντονο ενδιαφέρον. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρο. Είδατε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι Ιρλανδοί φίλοι. Και οι αποφάσεις που ελήφθησαν τις τελευταίες μέρες από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας οδήγησαν το δημόσιο έλλειμμα της Ιρλανδίας στο 32% του ΑΕΠ. Σε ένα χρόνο. Ο στόχος είναι να επανέλθουν στο 3% το 2014. Μου προκαλεί ρίγη αυτή η απόφαση. Φανταστείτε όμως την κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε τη στιγμή της συνδιαλλαγής με, τη... με το Συμβούλιο Υπεύθυνο για θέματα προϋπολογισμού για τον προϋπολογισμό του 2011. Δεν φαντάζομαι ότι δηλαδή μπορεί να χρηματοδοτήσει, μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κατά 2, 3, 4%. Ξανά η Μπάρμπαρα. Έχω σχεδόν, ε, το έχω πάρει μονότερμα. Έκανα ένα λάθο πριν. Για την περίπτωση τη Ιρλανδίας, που θα ψηφίσουμε στι 26 Οκτωβρίου, η <laughs> προθεσμία είναι 15 Οκτωβρίου για τις τροπολογίες. Έτσι είχα κάνει λάθο. 15 Οκτωβρίου, 10 η ώρα, είναι η καταληκτική προθεσμία, ούτω ώστε να μπορέσουμε να μεταφράσουμε τις τροπολογίες και σε όλες τις γλώσσες. Το 8, 9, 10, 11 το κάναμε, το 6 το αναβάλουμε, όπως σας είπα προηγουμένως. Έχουμε το σημείο 7, διορθωτικό προπολογισμό, αριθμός 6. Ο κύριος Γκουαλτιέρη δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σουριάν μπορεί να μας το παρουσιάσει. Το σημείο 6. Παρακαλώ κύριε Σουριάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορώ να εκφραστώ εξ ονόματος του συνεισηγητού μου και προτείνω να εγκριθεί χωρίς καμιά αλλαγή από την Επιτροπή μας η διόρθωση αυτή του προϋπολογισμού ο διορθωτικός προϋπολογισμός μάλλον. Διότι περί τίνος πρόκειται. Περί πρόκειται. Η δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων δεν είναι κάτι ουδέτερο, αλλά αυτό το ξέραμε, το ξέραμε. Και τώρα βλέπουμε ότι πράγματι απαιτείται παραπάνω, μεγαλύτερα απαιτούνται παραπάνω κονδύλια. είχαμε συμφωνήσει τον Απρίλιο να αρχίσει να λειτουργεί, τώρα θα λέμε ίσως τον Νοέμβριο ίσως. Η διόρθωση 6 λοιπόν βασίζεται στην ιδέα ότι θα υπάρξει μια τουλάχιστον τρίμηνη λειτουργία της υπηρεσίας για τους οποίους πρέπει να διασφαλίσουμε κονδύλια. Τώρα μας μιλάνε για δύο μήνες, δύο μήνες. Θεωρητικά λοιπόν τίθεται το ερώτημα. Τίθεται. Μήπως πρέπει να περικόψουμε το 1 τρίτο των προβλεπωμένων κοντιλίων. Ο Ζυγητής διαφωνεί. Θεωρεί ότι θα ήταν επικίνδυνο κάτι τέτοιο. Το Συμβούλιο δέχτηκε αυτή την περικοπή αλλά αν εμείς την απορρίψουμε θα χρειαστεί συνδιαλλαγή ταυτόχρονα με την μεγάλη συνδιαλλαγή. Άρα ούτε το Νοέμβριο θα μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί αυτή η υπηρεσία. Επομένως το μικρότερο κακό θα ήταν να διασφαλίσουμε τα ποσά ούτως ή άλλως. Καλύτερο είναι αυτό παρά να δοθεί αρνητική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν νομίζω ότι πρόκειται να υπάρξει καμία σοβαρή υπερδαπάνηση. Αν όμως παρελπίδα συνέβαινε κάτι τέτοιο μπορεί πάντα η Κομισιόν να προτείνει και άλλες μεταφορές. Με τον γνωστό τρόπο δεν γίνεται βέβαια διότι εδώ πρόκειται για ειδική θέση του προϋπολογισμού και δεν μπορεί να γίνει εκεί μεταφορά. Άρα, σύγχρονα συντομεύω, Πιστεύω ότι η πρόταση ως έχει πρέπει να εγκριθεί για να δείξουμε και την καλή μας θέληση προς τους εταίρους μας. Βέβαια θα χρειαστεί να τα ξαναδούμε όλα αυτά πολλές φορές. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι πρόκειται για διορθωτικό προπολογισμό 2010 για την ε, λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων για το τέλος του 2010 μόνο. Και οι τροπολογίες που θα ψηφίσουμε αύριο για να μπει στο αποθεματικό ένα τμήμα του προϋπολογισμού της υπηρεσίας αυτής αφορούν το 2011. 11. Ο Γκέβαν. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος μεταφέρω τη συγγνώμη του κ. Γουαλτιέρη, ο οποίος απουσιάζει για κάποιους λόγους, αλλά μου είπε να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο είπε ο Λάσλος Σουριάν, πως υπάρχει συμφωνία, πως πρέπει να υιοθετηθεί αυτό χωρίς τροπολογία, καθώς αποτελεί μέλος του πακέτου που πρέπει να συμφωνηθεί τον Οκτώβριο. Οπότε για εμάς δεν υπάρχει πρόβλημα να υιοθετηθεί. Ευχαριστώ Γέραν, ο κύριος Πόρτας. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ. Και εγώ έχω ένα ερώτημα προς τον κύριο Σούριαν. Δεν κατάλαβα καλά. Από ό,τι κατάλαβα ή από ό,τι άκουσα, η υπηρεσία αυτή θα ξεκινήσει να λειτουργεί τον ε, Νοέμβρη. Οπότε πρέπει να... Βλέπω εδώ πέρα πρέπει να εγγράψουμε τρεις μήνες και όχι δύο μήνες. Δεν υπάρχει κάποιος ε, κίνδυνος ε, εδώ πέρα. Μήπως δώσουμε παραπάνω χρήματα που υπάρξει. Έτσι. Πώς ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Ο Νομίζω πως η διερμηνία ήταν σωστή. Πράγματι, έχουμε τρεις μήνες προβλέψει ως στήριξη και δύο μήνες απαιτήσεων. Οπότε, θεωρητικά, θα υπάρχει δυνατότητα να κόψουμε κάτι. Αλλά για διαδικαστικούς λόγους, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα κάποια καθυστέρηση. Και η καθυστέρηση αυτή είναι αντίθετη με τις συμφωνίες. Οπότε, δημοσιονομικά σκεπτόμενοι, είναι λογικό να κόψουμε, αλλά υπάρχουν και άλλα συμφέροντα εδώ πέρα. Και δεδομένου του ότι δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό, προτείνω να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ πέρα. Γιατί τώρα είναι τρεις αυτό είναι το ερώτημά σας. Γιατί όταν είχαν προετοιμάσει τον ε, τροποποιητικό προπλογισμό υποθέταν πως θα είχαμε τρεις μήνες. Και τώρα βεβαίως ε, βλέπουμε πως ε, θα το συζητάμε και θα το αλλάζουμε και θα μιλάμε για ένα μήνα. Και είναι βεβαίως ένα ζήτημα εξωπρέπειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαντάει στο ερώτημα του Κίσιγκερ σε ποιον να τηλεφωνήσω. Ή εν μέρη απαντάει. Ευχαριστώ κύριε Σαρθό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις που τις ήθελα για αύριο βέβαια να τις κάνω, αλλά μια που το συζητήσαμε η κυρία Άστον είπε πως ολόκληρη υπηρεσία, ολόκληρη υπηρεσία δεν θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό και μιλάμε τώρα εδώ πέρα για άλλα 18 εκατομμύρια που ζητούν για τις επιπλέον θέσεις. Άρα, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν βεβαίως και οι ψηφοφόροι μου στην Ολλανδία. Η, ουδετερότητα του προπολογισμού πρέπει να λάβει υπόψη και τους 28 προϋπολογισμούς, τους 27 εθνικούς και τον 28 τον ευρωπαϊκό. Το παλάτι, λοιπόν είναι στο στρατόπεδο των ε, κρατών μελών. Αυτό λέω και στην κυβέρνηση μου στη Γαλλία. Υπάρχουν δύο τρόποι να δημιουργήσουμε αυτή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ο ένας τρόπος λέει, έχουμε 27 εθνικές διπλωματίες, θα έχουμε και μια 28η. Αν αυτή είναι η προκρινόμενη λύση, νομίζω ότι είναι λάθος και από γραφειοκρατική άποψη και από διπλωματική και από οικονομική. Υπάρχει όμως ένας άλλος τρόπος. Θα ασχοληθούμε με κάποια μεγάλα διπλωματικά θέματα, όχι πια σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό. Και θα μεταφέρουμε ε, εθνικούς πόρους στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να ασχοληθεί με αυτά. Αν επιλέξουμε αυτή τη λύση, όχι μόνο δεν θα υπάρξει αύξηση του άχθους για το φορολογούμενο, δεν θα υπάρξει αύξηση των δημοσίων δαπανών, αλλά θα υπάρξει και μείωση. Γιατί αν σε 10, 15, 20 χρόνια έχουμε μία μόνο ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία για 27 κράτη-μέλη, θα κάνουμε τρομακτικές οικονομίες. Και αυτό είναι πολιτική επιλογή, έτσι. Σε ό,τι αφορά την ουδετερότητα, τα 18 εκατομμύρια που προσθέτονται εδώ, που του χρόνου θα φτάσουν σε 34 εκατομμύρια. Πρόκειται για μεταφορά δαπανών ουσιαστικά του Συμβουλίου ή των κρατών μελών ή της Κομισιόν προς την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και επομένως η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα χρειαστεί επιπλέον μέσα, γιατί δημιουργούμε μια υπηρεσία που δεν υπήρχε μέχρι τούδε και που έχει και τη δική του θέση στον προπολογισμό, τη θέση υπαριθμών 10. Αλλά έχετε πολύ δίκιο που λέτε όλοι ότι πρέπει να προσέξουμε ότι σε ένα ή δύο χρόνια πρέπει να φτάσουμε σε ένα πλατό και να μην προχωρήσουμε παραπάνω. Και το λέω και για τον επόμενο εισηγητή, του επόμενου προπολογισμού του, του 2012 και 2013. Θα πρέπει να δούμε τι οικονομίες γίνονται στα άλλα θεσμικά όργανα και στα κράτη-μέλη ως αντιστάθμιση για αυτή την αύξηση σε πόρους σε προσωπικό, σε πιστώσεις λειτουργίας και σε επιχειρησιακές πιστώσεις που θα πρέπει να αυξηθούν, που θα δώσουμε στην Άστον και στην υπηρεσία της. Ποια είναι αυτή η αντιστάθμιση λοιπόν που γίνεται, αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν, θα, δεν το λόγο, θα ψηφίσουμε αύριο. Μου λένε ότι υπάρχουν πέντε τροπολογίες από την κυρία Γκρέσλα που μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα υπάρχουν σήμερα το βράδυ ελπίζω σε όλες τις γλώσσες, ούτως ώστε κάθε ομάδα να προετοιμάσει την ψηφοφορία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο στα αγγλικά. Που είναι η μητρική γλώσσα της κυρίας Γκρέσλε βέβαια, έτσι. Ειδικά για τα δημοσιονομικά είναι τα αγγλικά. Αραβικά νούμερα είναι αυτά. Ούτως ή άλλως. Θα τα ψηφίσουμε όλα αυτά αύριο λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Αυτό ήταν το σημείο 7. Και τώρα πάμε στις μεταφορές, σημείο 12. Αλλά αύριο είναι ψηφοφορία. Αυτό είναι... Θα το συζητήσουμε αύριο. Αφορά την ψηφοφορία. Κύριε Σούριαν. Έχουμε 7 μεταφορές κονδυλίων να ψηφίσουμε, πιστώσεων να ψηφίσουμε αύριο. Έτσι δεν είναι κύριε Σουριάν. Οι τέσσερις πρώτες αφορούν το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, μόλις τη συζητήσαμε και θα τη ψηφίσουμε αύριο. Έπειτα, για τα άλλα θεσμικά όργανα, έχουμε κάποιες μεταφορές πιστώσεων, επίσης. Ο κ. Μάνκα δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω. Η σοσιαλιστική ομάδα Μπορεί να μας πει αν κάποιος μπορεί να αντικαταστήσει τον κύριο Μάνκα ή... το να τον αντικαταστήσω εγώ. Αν δεν είναι εδώ θα είμαι εγώ εκπρόσωπος του εισηγητή. Εντάξει. Αυτό είναι το σημείο 13. Πολύ ωραία. Σημείο 14, 15, 16, 17. Τίποτα δεν έχουμε να πούμε για αυτά. Κλείσαμε, τελειώσαμε την ημερήσια διάταξη. Κλείνω εδώ τη συνεδρίαση και θα κρατήσω τους συντονιστές και τις, και και τους συντονιστές. Να παραμείνουν οι διερμηνείς παρακαλώ, θα συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά με τη συνεδρίες των συντονιστών.